Välkomna Καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή τη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Vivian Ρέντινγκ. Καλώς ήρθατε σε αυτή την Επιτροπή. Η κυρία Ρέντινγκ είναι αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης επίτροπο δικαιοσύνη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ηθαγένεια. Και τα θέματα που θα συζητήσουμε με την κυρία Ρέντινγκ σήμερα το απόγευμα είναι μελλοντική στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Όπω γνωρίσουμε αυτό καλύπτει έναν ευρύ τομέα πολιτικό. Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία αυτή να μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με την Επίτροπο. Δηλαδή τη μελλοντική στρατηγική για την ισότητα των Φίλων. Σας καλωσορίζουμε ένθερμα και θα σας δώσω κατευθείαν το λόγο, κυρία Ρέντινγκ. Thank you, Madam Chair. And hello, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Γνωρίζετε ότι μία από τις πρώτες δράσεις της νέας Κομισιόν ήταν η θέτηση της χάρτας των γυναικών και κάθε ένας επίτροπος αλλά και η Κομισιόν στο σύνολό της ανέλαβαν δέσμευση ότι κατά τη διάρκεια των πέντε αυτών ετών θα αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και ότι θα θέσουμε ως προτεραιότητα το θέμα αυτό και θα καταπολεμήσουμε φυσικά και την παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμα το οποίο εντοπίζει προσδιορίζει μια σειρά δράσεων για να σημειώσουμε πρόοδο για την ισότητα των δύο φίλων. Η κυρία Φιγκερέιτο ήταν πραγματικά μεγάλη πηγή έμπνευση. Όπως σας είπα, Καλή είναι θεωρία, όμως πρέπει να ακολουθείτε και με πράξεις. Και ακριβώς αυτό τώρα προετοιμάζουμε. Δρομολογείται η Κομισιόν. Εργάζεται επί της στρατηγικής, η οποία θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο, Πρόεδρε. Έτσι λοιπόν μπορείτε ήδη να σχεδιάσετε το έργο της δικής σας Επιτροπής βάσει αυτής της στρατηγικής. Και όπως σας είπα, αυτή η στρατηγική δεν θα είναι μόνο η στρατηγική της ε, Επιτρόπου που είναι αρμόδια για τις ε, γυναίκες, αλλά θα είναι στρατηγική ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό κάλεσα και τους ε, συναδέλφους, τους υπόλοιπους επιτρόπους γραπτός να προτείνουν δράσεις στο δικό τους τομέα, στα δικά τους χαρτοφυλάκια, προκειμένου να καταστήσουν την ισότητα των δύο φύλων αυτό στόχο στα χαρτοφυλακιά τους και φυσικά αυτό θα προσαρμοστεί στη στρατηγική. Έτσι λοιπόν, όλοι εσείς αποσχολείστε και με άλλους τομείς της πολιτικής, μπορείτε να συζητήσετε στα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα με τους αρμόδιους επιτρόπους. Όπως ε, αναγραφόταν και στη χάρτα, η στρατηγική θα βασίζεται σε πέντε προτεραιότητες την οικονομική ανεξαρτησία, ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία, ισότιμη πληρωμή για ε, ισότιμη εργασία και εργασία ισότιμη αξία, ισότητα, στη λήψη αποφάσεων, αξιοπρέπεια και αιρεότητα και τεθεί τέλο στην ε, βία κατά των γυναικών και ισότητα των δύο φύλων εκτός της Ένωσης. Δεν είμαι ακόμη σίγουρη, αλλά ίσως αυτά Μπορεί να προσθέσω και ένα διατομιακό κεφάλαιο που θα διερευνά το ρόλο των φίλων, την νομοθεσία και τα εργαλεία διακυβέρνηση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και ένα έκτο κεφάλαιο που θα προσθεθεί. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες από αυτού. Σε ό,τι αφορά την οικονομική εξαρτησία και για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης το 2020, Ξέρω ότι σε αυτή την Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια εσείς έχετε συζητήσει το θέμα αυτό. Ο στόχο ε, του 75% του στόχου του ποσοστού 75% απασχόληση για άντρες και γυναίκες μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν απασχολούνται περισσότερες γυναίκες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά εργασίας και στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αλλά Φυσικά δεν αρκεί το να έχουν πρόσβαση οι γυναίκε στι θέσει εργασία, αλλά πρέπει να δούμε και ποια είναι η ποιότητα των θέσεων εργασία αυτών όπου απασχολούνται οι γυναίκε. Και δεν χρειάζεται να σα το πω αυτό, το γνωρίζετε. Οι γυναίκε ε, εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται σε επισφαλεί θέσει εργασία ε, και σε ήμια απασχόληση. Όμω, Φυσικά η οικονομική ανεξαρτησία δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς να υπάρχουν ε, αυθεντικές ευκαιρίες για τη συμφιλίωση της επαγγελματική με την ιδιωτική ζωή. Και εδώ πραγματικά στα περισσοτερα κρατημέλη πρέπει να υπάρχει περαιτέρω υποστήριξη για να έχουμε διευθετήσεις ε, για ευέλικτη εργασία και φυσικά να έχουμε και εγκαταστάσεις φροντίδας για τα παιδιά. Και ε, για τους υπόλοιπους εξαρτώμενους, όταν αναφέρομαι στους υπόλοιπα εξαρτώμενα άτομα, αναφέρομαι στο πρόβλημα της γύρασης του πληθυσμού. Ξέρετε, ε, Πρόεδρε, στο εγγύς μέλλον θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο ελληνικής μεταξύ των γενναίων. Αυτό αποτελεί τη βάση της λειτουργίας των κοινωνιών μας εδώ στην Ευρώπη. Και φυσικά οι γυναίκες διαδραματίζουν ειδικό ρόλο εδώ. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι που θα το επιλύσουμε αύριο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αρχίσουμε να το εξετάζουμε τώρα, έτσι ώστε τα επόμενα έτη να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Γιατί η φροντίδα των ηλικιωμένων κυρίως ήταν στα χέρια των γυναικών μέχρι σήμερα. Και μιλάμε για πολλές γυναίκες οι οποίες δεν απασχολούνταν επαγγελματικά. Φυσικά όλα αυτά όμως θα αλλάξουν. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες αυτό το θέμα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, αλλά πολλές φορές ε, και παράλληλα πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αλλά και επειδή οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες, θα καταστεί ένα γυναικείο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, τι θα κάνουμε με την αλληλεγγύη και την της ισορροπίας. Είναι μια ερώτηση αυτή, ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όχι τώρα αμέσω, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και να δούμε τι μπορούμε να προετοιμάσουμε. Τώρα, η γεφύρωση του κενού στους μισθούς μεταξύ των δύο φύλων. Εδώ σχεδιάζουμε την ανάληψη πολιτικών σε συνεργασία με τους κοινωνικούς αδέρφους και τις εταιρείε και μας αρέσει η ιδέα για να έχουμε αυτή την ημέρα της ε, ισότιμης αμοιβή και να προκαλέσουμε συζήτηση και να ασχοληθούν και τα ΜΜΕ ε, με αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν θα η πρόταση αυτή. Ισότητα στη λήψη αποφάσεων. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ε, είναι κάτι που ισχύει και πρέπει να αναλάβουμε δράση για να αλλάξουμε τις νοοτροπίες προκειμένου να σημειωθεί η πρόοδος. Δεν αποκλείω τη δυνατότητα να προωθήσουμε νομοθεσία στον τομέα αυτό. Ένα από τα κύρια, από τα σημαντικά θέματα στην ατζέντα μας, στη στρατηγική μας, είναι αποφασιστική δράση για να κατολμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και να διασφαλίσουμε ότι τα θύματα προστατεύονται αποτελεσματικά όπως ήδη ανακοίνωσα, εργάζομαι επί ενός ε, συνολικού πακέτου για τα θύματα και θα το παρουσιάσω το πρώτο ήμιση του 2011. Επίσης, αναλαμβάνουμε δράση για να εξελίψουμε τον ακριτηρισμό των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες και Τώρα εξετάζω μέτρα που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και μέτρα ποινικού δικαίου αν χρειαστεί και πιθανότητα θα χρειαστεί γιατί δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να ανεχόμαστε μια τέτοια βίαιη πρακτική. Καμία δικαιολογία και φυσικά αν κάνουμε κάτι στην Ευρώπη για τον ακριτηρισμό των γεννητικών οργάνων αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μιλήσουμε με μια νέα φωνή και υιοθετήσουμε και μια κοινή λογική στις εξωτερικές μας σχέσεις. Εδώ θα προτείνουμε καταρχήν να διασφαλίσουμε ότι οι υποψήφιε προσέγγιση χώρα θα σέβονται πλήρω την ομοθεσία μα. Και δεύτερον, θα συνεργαστούμε με του εταίρου μα και με τα κράτη αλλά και με κρατικού παράγοντε για να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων. Και είμαι πάρα πολύ θετική σε σχέση με τα μέτρα που θα λάβουν οι συνάδελφοι στους τομείς της αναπτυξιακής βοήθειας, ε, παραδείγματος χάρη, γιατί τους απασχολούν πάρα πολύ και τα θέματα των γυναικών. Κάθε χρόνο η έκθεση της Επιτροπής ε, για την πρόοδο που έχει υλοποιηθεί και για τις προκλήσεις που παραμένουν στον τομέα της ισότητας των φύλων θα παράσχουν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο τη βάση για έναν αιτήσιο ε, διάλογο υψηλού διαλόγου και με άλλους κύριους πρωταγωνιστές, όπως προτείνετε εσείς, Πρόεδρε. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας και να καταστήσω την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο εξωτερικό. Και μια πληροφορία. Γνωρίζετε ότι από την 1η Ιουλίου και μετά έχουμε το Γενικό Διευθυντήριο της Κομισιόν για τη Δικαιοσύνη ανεξάρτητο. Έχουμε διχωριστεί από τις εσωτερικές υποθέσεις. Έχουμε τη διεύθυνση αυτή για τη δικαιοσύνη λοιπόν. Και μια γυναίκα είναι γενική διευθύντρια, η κυρία Φρανσός Λεμπάη. Γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες με τα κατάλληλα προσόντα, απλώς πρέπει κάποιος να τις βρει και να τις βάλει σωστή θέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είμαι πεπισμένη ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, όπως και εγώ, συμφωνούν ότι οι γυναίκε με προσόντα υπάρχουν αρκεί να βρεθούν στην κατάλληλη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγική σα ομιλία. Περιμένω με ανυπομονησία την συζήτηση. Πρώτη θα λάβει τον λόγο ή μάλλον Πρώτο, ο κύριο Ρωμέβα. Έχει το λόγο κύριε Ρωμέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ και που είστε εδώ αλλά και για τα όσα είπατε και τα σχόλιά σας. Το δικό μου σχόλιο αναφέρεται περισσότερο σε δύο προσθήκες ή δύο, μια παράκληση μάλλον να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες. Αφενός για την εκτίμηση που εγκρίναμε στο κοινοβολίο σχετικά με ε, ομοφιλόφιλους που για μας είναι πάρα πολύ το θέμα είπαμε συγκεκριμένα ότι στον οδικό χάρτη πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των προσώπων αυτών. Ζητήσαμε να περιληφθούν όχι μόνο οι πολλαπλές διακρίσεις και αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο, διότι ορισμένες ε, χώρες μέλη προβάλλουν τις χέρειες, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ζητήσαμε να γίνει διαβούλευση με ειδικέ οργανώσεις για θέματα ισότητα των φύλων, να γίνει μια εκστρασία ευαισθητοποίηση ε, για ε, ανθρώπους που έχουν αλλάξει φύλλο και που για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρομαι στη νέα στρατηγική για την ισότητα των φίλων, η οποία θα πρέπει αρρητά ε, να ε, περιλάβει και θέματα αλλαγής φύλου. Για τον Σεπτέμβρη, για το φθινόπωρο δηλαδή, σχεδιάζουμε ακρόαση μαζί με την συνάδελφό μου Κορνέλησεν για το θέμα αυτό και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για το θέμα αυτό. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για το θέμα αυτό και σας υποσχόμαστε την υποστήριξη όχι μόνο τη παρούσα επιτροπή αλλά και του Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα αναλάβετε προ την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερη σύντομη ερώτηση Βλέπω και δύο συναδέλφους μου ε, που θα μπορούν να πούν περισσότερα νομίζω γιατί έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Θέλω να το αναφέρω εν πάση περιπτώσει. Σε σχέση με το European Protection Order που είναι σημαντικό θέμα και ευαίσθητο. Και τα πράγματα μέχρι τώρα είναι περίπλοκα. Αλλά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλοί από εμά υποστηρίζουμε απολύτως την πρωτοβουλία αυτή διότι θεωρούμε ότι την χρειαζόμαστε στην πράξη το καλύτερο είναι, σύμφωνα βέβαια με την νομική βάση, αλλά να είστε βεβαία ότι η θέληση της πλειοψηφίας, την οποία εκτιμώ εγώ ως πλειοψηφία, αν και δεν έχουμε ψηφίσει ακόμη, πάντως πολλοί από εμά την υποστηρίζουμε και παρακαλούμε να αναλυθεί κάποια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας υποβληθεί κάποια βάση για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμέβα. Πριν δώσω τον λόγο στο επόμενο πρόσωπο που έχει εγγραφεί, θα σας πω μόνο ότι υπάρχουν 11 εγγεγραμμένοι. Παρακαλώ όλες και όλους να δείξετε αλληλεγγύη μεταξύ σας. Να σκεφτείτε και όλους και όλες εκείνους που θέλουν ακόμη να λάβουν το λόγο Πέστε ό,τι θέλετε να πείτε βεβαίως, αλλά με συντομία, για να αφήσουμε χρόνο στην Επίτροπο να απαντήσει. Άρα, παρακαλώ, το δυνατόν συντομότερη. Η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ, κύριε Ρέτινγκ, που ήρθατε. Απίλαυσα την συζήτησή μας προμηνώς στο Στρασβούργο και περιμένουμε ανυπομονησία την επόμενη. Το κεφάλαιο που αναφέρατε για την ε, ισότητα των φύλων ε, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Είπατε ότι ίσως προτείνεται νομοθεσία για θέματα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έχουμε κάνει κάθε άλλη δυνατή προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες και δεν πήγαν πολύ καλά οι προσπάθειες αυτές. Δεν άκουσα να λέτε και θα ήθελα να μου απαντήσετε. Πρώτα-πρώτα για την πατρική άδεια. Αρχίζω και λέω τα ίδια και τα ίδια. Αν θέλουμε όμως περισσότερες γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας, πρέπει η φροντίδα των παιδιών να κατανεμηθεί καλύτερα μεταξύ των φίλων και να δοθεί ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα στους άνδρες ότι ε, καλούνται και αυτοί να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για τη φροντίδα των εξαρτώμενων προσώπων, εάν θέλουν ε, να υπάρχει αυτή η ισότητα. Είπατε επίσης για την δέσμευση ολόκληρης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι οι υπόλοιποι επίτροποι θα υποβάλουν και αυτοί οι σχέδια προς την κατεύθυνση αυτή. Πώς θα παρακολουθείτε αυτό το έργο, ωστόσο, στην εξέλιξή του. Η Επιτροπή Απασχόλησης ασχολείται με τις Employment Guidelines και έχουμε βάλει και μια σημαντική διάσταση ισότητας φύλων. Η Κομισιόν θα αναλάβει δράση να το προωθήσει το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο. Το ίδιο για το πράσινο βιβλίο για τις συντάξεις. Έχει και, υπάρχει και εδώ μια ισχυρή διάσταση ισότητας φύλων που πρέπει να ε, τονιστεί. Στις διαπραγματεύσεις για το EEAS περιλήφθηκε μια διάταξη για την εξασφάλιση σε όλα τα επίπεδα της ισότητας των φύλων. Πρέπει να γίνει πολύ ε, ξεκάθαρη παρακολούθηση, monitoring, monitoring δηλαδή, ώστε από την αρχή να υλοποιείται και θα ήθελα να μου πείτε η δική σας εμπλοκή ποια θα είναι. Ευχαριστώ κύριε Κορνέλισε. Κύριε Μπάουερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να χαιρετήσω αυτή τη δυνατότητα που μας δίνεται να κάνουμε μια συζήτηση με την ε, κυρία Επίτροπο ε, για κάποια πολύ επίκαιρα θέματα. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της ε, Οδηγία ε, για την ε, άδεια και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας ε, θέση σε ό,τι αφορά την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Ε, μελέτη αξιολόγησης που θα αξιολογηθεί, ελπίζουμε, στο δικής μέλλον. Αλλά όταν είχαμε αποφασίσει να εκπονηθεί αυτή, εκείνη η μελέτη, μας είχατε υποσχεθεί ότι θα μας ότι θα αναλάβετε κι εσείς ένα κομμάτι αυτής της ευθύνης, ας το πούμε έτσι, και είχατε δεσμευτεί ότι θα εκπονήσετε μια μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου για την άδεια πατρότητα. Ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το κόστος, ε, το κόστος ε, το οποίο θα προκύψει μέσα από, αυτή την, ε, από αυτές τις άδειες ε, και ούτω καθεξής. Και τώρα ενημερωθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η δική σας ε, αξιολόγηση αδικτύπου θα είναι έτοιμη του χρόνου. Άρα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Θα υπάρξει μια δήλωση από τη δική σας πλευρά σε ό,τι αφορά την ε, μελέτη αντικτύπου. ίσως θα έπρεπε να ξανανοίξουμε εκείνη τη συζήτηση ε, που έλεγε ότι θα πρέπει να έχουμε τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας σε ό,τι αφορά την ε, άδεια μητρότητα σε μια οδηγία και όλα τα υπόλοιπα σε κάτι άλλο. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την άδεια μεταποδοχών, ε, ε, πώς ε, θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να παράσχετε κάποια κίνητρα, γιατί είδαμε ότι σε πολλές χώρε υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωση, γιατί δεν υπάρχει και μια δημοσίευση ό,τι αφορά, δεν, δεν λαμβάνει δημοσιότητα το ζήτημα τη ε, μισθολογικής διαφοράς μεταξύ άντρων και γυναικών. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της αύξησης της απασχόλησης των γυναικών. Ε, ακούσαμε ότι γύρω στο 1 τέταρτο των απασχολούμενων γυναίκες. Οπότε ε, ε, θεωρούμε πως εάν δεν συμφιλώσουμε κατά κάποιο τρόπο την οικογενειακή ζωή με την απασχόληση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αλλάξουμε αυτό το ποσοστό. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε ε, σκοπό να θέσετε ε, κάποιους μικρούς ε, στόχους βαρκελώνης εντό εισαγωγικών σε ό,τι αφορά την παιδική φροντίδα. Γιατί όπως θα θυμόσαστε οι τελευταίοι στόχοι της Βαρκελόνης δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν. Ποια λοιπόν θα είναι τα βήματά σας, ποιος ο στόχος σας σε αυτό το τομέα και σας ευχαριστώ και το προτείνω για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ευχαριστώ γεγονό ότι έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψε μαζί σα, γιατί ε, απαντάτε με πολύ σαφή τρόπο στα ερωτήματά μα ε, και επιδεικνύεται μεγάλη δέσμευση ό,τι αφορά τι ε, προτεραιότητε που θέλετε. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη δημογραφικού χαρακτήρα κρίση, τι ακριβώ σκοπεύετε να κάνετε ω προ τον αντίκτυπο τη δημογραφική σύγκριση στι γυναίκε ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά ε, το σχέδιο καταπολέμησης ε, της, ε, της δημογραφικής κρίσης, με βάση μια πρόσφατη διάσκεψη διαπιστώσαμε ότι το 80% της φροντίδας παρέχεται, δηλαδή σε ό,τι αφορά την οικογένεια, από την ίδια την οικογένεια και το 90% από τις γυναίκες. Επίσης, το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το γεγονό ότι πολλέ φορέ καλούμαστε να λάβουμε κάποιε αποφάσει, αλλά δεν έχουμε κατάλληλη ενημέρωση, δεν έχουμε τα κατάλληλα δεδομένα από το κοινωνικό τομέα. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω εάν έχετε σκοπό να χρηματοδοτήσετε κάποια πιλωτικά προγράμματα ή κάποιε μελέτε οι οποίε θα μα δώσουν τη δυνατότητα να είμαστε πιο επαγγελματίε σε ό,τι αφορά την ε, άσκηση τη πολιτική μα. Σα ευχαριστώ. Ehm, ευχαριστώ. Κύριε Ρομέρο και μετά θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία στην Επίτροπο να απαντήσει πρώτα. Κύριε Ρωμήρο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ραντίνκ που παρευρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και επίσης ε, σας ευχαριστούμε και για την προσωπική σας διαδρομή για την υπεράσπιση των γυναικών αλλά και για την ε, πρωτοβουλία που αναλάβατε για την ε, νομοθεσία περί διαζυγίων. Μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή και γι' αυτό θα ήθελα ένθερμα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι η συγγήτρια για την έντολη ε, προστασία ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις για αυτή την πρωτοβουλία των κρατών μελών η συζήτηση για την οποία ξεκίνησε κατά την Ισπανική Προεδρία δεν υπάρχει μια οδηγία για τη βία, γιατί μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και όχι για διεθνή ε, εγκλήματα, αδικήματα, αλλά μετά την ε, υιοθέτηση της συνθήκης Λισαβόνας και της χάρτας των δικαιωμάτων θα έπρεπε να σκεφτούμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα ως βάση για τις οδηγίες. Τώρα ίσως ανοίγεται ε, ένα νέο πεδίο, αλλά πραγματικά υπάρχουν ε, εγκλήματα που, και αδικήματα που θίγουν ε, την, την φυσική ακυρεότητα των γυναικών. Και αυτό φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις για την εντολή προστασία και ελπίζω να μπορέσετε να απαντήσετε και να τις διασκεδάσετε. Η Κομισιόν δεν μας παρουσίασε κανένα επίσημο έγγραφο, αλλά ενίοτε γίνεται λόγος για την πρωτοβουλία αυτή ότι ουσιαστικά θα μπορέσει να καλυφθεί σε δύο στάδια. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται η Κομισιόν τα μιλά για δύο στάδια και θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης τι πιστεύετε για το ότι ε, τα κράτη-μέλη μιλούν για μια αρχή που διορίζεται στα διάφορα κράτη για να αποφασίσει για ε, το ποιο δικαστήριο είναι το αρμόδιο όταν εκδίδεται μια ΕΠΟ μια τέτοια εντολή προστασία. Έτσι λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω πώ σας φαίνεται σα αυτή η δυνατότητα να υπάρχει μια αρχή που έχει επιλεχθεί σε κάθε κράτο μέλο για να αποφασίζει την δικαιοδοσία. Όπως ε, ξέρετε, αν ε, τα ασφαλιστικά μέτρα σε κάποιες χώρες είναι διοικητικού χαρακτήρα ή αστικού χαρακτήρα, σε άλλες χώρες ε, είναι είτε ποινικού χαρακτήρα ή στη δική μου χώρα έχουμε συγκεκριμένα δικαστήρια που δικάζουν υποθέσεις οικογενειακής βίας. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο ένα μέτρο να μπορέσει να καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις διαφορές ε, των ε, διάφορων νομικών συστημάτων και των νομικών παραδόσεων. Έτσι λοιπόν, Τώρα να έχουμε μία αρχή ε, τέτοιου είδους ε, η οποία θα διορίζεται ε, για να καθορίσει το αρμόδιο δικαστήριο θεωρήσαμε ότι ίσως να αποτελούσε μία λύση. Θέλουμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Φυσικά είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα πέρα από νομικό. Αλλά όπως είπε και ο συντηρητικός πρόεδρος της Σουηδίας το νομικό πρόβλημα πρέπει να το λύσουν οι νομικοί. Εμείς είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εσείς ε, και εμείς εδώ είμαστε και πολιτικοί αλλά και προσωπούμε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε μόνο για ένα πρόβλημα βίας όταν αυτό έχει να κάνει με τους εξαναγκαστικούς γάμους ή ε, με την ε, κλιτερδεκτομή. Έτσι λοιπόν πρέπει να μιλάμε και για την βία κατά των γυναικών που λαμβάνει χώρα σε κάποιες χώρες ε, δυστυχώς και μιλάμε για χώρες ε, όπου αυτοί που διαπράττουν τη βία είναι πραγματικά οι πολίτες μας. Έτσι λοιπόν ε, στις 4 ε, Ιουνίου όταν συνεδρίασε το Συμβούλιο ΔΕΗ ε, μία δημοσιογράφος εδώ στις Βρυξέλλες, μία δημοσιογράφος από τη Βουλγαρία, η κυρία Παρασκευό δολοφονήθηκε και ο σύντροφ, αυτός που παρουσιάστηκε ως σύντροφός της κατήγγειλε το συμβάν στο Λουξεμβούργο. Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε και με ποιο τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα και πάλι το λόγο στην Επίτροπο Ρέντινγκ για να δώσω κάποιες πρώτες ε, Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν απαντώντας τον κύριο Ρωμαβά. Ε, συμφωνώ ότι το ζήτημα της ε, πολλαπλής διακριτικής ε, μεταχείρισης απέναντι δηλαδή σε διαφελικά άτομα ομοφυλόφιλους και ούτω καθεξής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και οι συνεργάτες μου ήταν, ήταν πάντοτε παρούσα όποτε γίνεται μια σχετική συζήτηση είτε εδώ είτε στα κράτη-μέλη για να δείξουμε ακριβώς ότι παίρνουμε στα σοβαρά αυτά τα ζητήματα ε, και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι κάνετε αυτή την ακρόαση για να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση ε, του ευρωστινού. Γνωρίζετε πως ε, όποτε έχει υπάρξει ένα πρόβλημα σε κάποιο κράτος μέλος εγώ έχω τοποθετηθεί. Προσπαθώ δηλαδή να ε, αμβλύνω λίγο αν θέλετε τις υπερβολικά ακραίες ε, θέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Το πρόβλημα λύνεται μέσω της ε, οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων του 2006. Εκτός τώρα του χώρου της απασχόλησης Όπω γνωρίζετε η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων έχει ε, μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και δεν ξέρω αν είπα εδώ σε αυτή την Επιτροπή, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, δεν υπάρχουν και πολλέ ελπίδε ότι θα ξεμπλοκάρει αυτή η οδηγία στο Συμβούλιο καθώ όπω γνωρίζετε χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο για να περάσει. Άρα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα διαφορετικά από το να προσπαθήσουμε απλά να ξεμπλοκάρουμε αυτή την οδηγία, τουλάχιστον προς το παρόν. Σε ό,τι αφορά την εντολή προστασία. Είναι ένα πολύ περιπλοκό ζήτημα και ακριβώς επειδή είναι ένα περιπλοκό ζήτημα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα νομικά ζητήματα που υπάρχουν εδώ. Ναι, εντάξει, τα νομικά ζητήματα απασχολούν τους ε, ε, νομικούς, αλλά εμείς είμαστε που θεσπίζουμε νόμους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, θεσπίζουμε, να παράγουμε νόμους με ε, τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίσουν νομική βεβαιότητα. Έτσι ώστε οι δικηγόροι και οι δικαστές απλώς να καλούνται να εφαρμόσουν αυτό το νόμο και όχι να αμφισβητούν, αν θέλετε, να εκατολογούν σε σχέση με το, με το νόμο. αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια τέτοια ρύθμιση των εντολών προστατευτικών μέτρων, ώστε εφόσον υπάρχει μια τέτοια εντολή σε ένα κράτο μέλο, να αναγνωρίζεται και σε άλλο κράτο μέλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί εδώ να κάνει μια διασυνοριακού χαρακτήρα δουλειά, βοηθούμενη και από τι προπαρασκευαστικέ εργασίε που έγιναν κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία. Και για να αποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Άννα είναι η Εθνική Ορτή της Γαλλίας. Σήμερα βιβλα Φρανς, τα Επίτροπος. Αύριο λοιπόν στις 15. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια δημόσια ακρόαση προκειμένου να εξεταστεί το συνολικό πακέτο των πρακτικών μέτρων το οποίο θα ε, παρουσιαστεί μέσα στο 2011 και θα καλύπτει τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των ε, θυμάτων εγκλήματος και βίας. Γενικά θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των γυναικών. Έτσι λοιπόν εδώ ξεκινάμε με συγκεκριμένο έργο το οποίο θα κάνουμε για να έχουμε και συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν νομική βεβαιότητα για τα θύματα. Τώρα, ε, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Κονέλης. Το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση και τη λήψη των αποφάσεων. Η νομοθεσία δηλαδή, την οποία προβλέπουμε, εδώ θα πρέπει να πω ότι δεν θα πρέπει να χρειαστούμε 5 ή 10 χρόνια μελετών προσπαθώντας να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα πρέπει να κινηθούμε σταδιακά, με βήματα, για να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Και όταν λέω τελικό στόχο, είναι να έχω τέλος την, την αρμοδιότητα. Ναι, ναι. σε ό,τι αφορά τώρα την άδεια πατρότητας που σχετίζεται και με άλλα ζητήματα που έθεσαν μεταξύ άλλων η κυρία Μπάουερ, σχέση για παράδειγμα μεταξύ πατρικής και μετρικής άδειας έδειας μητρότητας πατρότητας. Γνωρίζω πως έχει ξεκινήσει η ειδική αξιολόγηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως σας ε, ε, υποσχεθήκαμε υπάρχει μια μελέτη αντικτύπου από την πλευρά της Επιτροπής σε ό,τι αφορά το κόστος που θα προκύψει από την παράταση, από τη μεγαλύτερη δηλαδή περίοδο άδεια ε, μητρότητα, αλλά ε, και σε σχέση με την άδεια πατρότητας. Και πράγματι, ναι, χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για να μπορούμε να προβαίνουμε σε καλές μελέτες αντικτύπου. Δεν έχετε ε, ως κοινοβούλιο αυτή την εμπειρία και το Συμβούλιο δεν έχει αυτή την ε, εμπειρία των ε, μελετών αντικτύπου. Δηλαδή το Συμβούλιο προβαίνει σε μία πρόταση χωρίς να έχει κάνει καμία μελέτη και μετά έρχεται η μελέτη και ε, δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εμείς ως Επιτροπή είμαστε υποχρεωμένοι να εκπονούμε μελέτες αντικτύπου και αποτελούν μία υγιή, μία σταθερή βάση. Γιατί αν υπάρχει μία τέτοια μελέτη μπορεί κανείς να βασίσει σε πολύ πιο ε, σταθερά θεμέλια την νομοθετική πρόταση. Άρα λοιπόν καλό είναι μερικές φορές να παίρνουμε λίγο παραπάνω χρόνο να καθυστερούμε παραπάνω για να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών ε, οργάνων που είναι αρμόδια ως ε, νομοπαραγωγή και βέβαια για να βρεθεί και μια συμφωνία και με τους ενδιαφερόμενους. Και εδώ περνάω στο ερώτημα της κυρίας Μπάουερ Μήπω θα πρέπει να έχουμε δύο ξεχωριστές προτάσει. Αφενό άδεια και αφετέρου άδεια και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Σε ένα άλλο δηλαδή νομοθέτημα. Και ίσως αυτό πράγματι να έχει νόημα. Γιατί όπως βλέπετε και εσεί οι ίδιοι, εάν προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τα πάντα σε μία νομική πράξη, σε ένα πακέτο, ε, ενδεχομένως να καθυστερούμε όλη την όλη διαδικασία. Και έλαβα, δεν ξέρω, ε, τις τελευταίες μέρες, πριν από μια εβδομάδα, από τη Συνομοσπονδία, την Εμπορική Συνομοσπονδία την Ευρωπαϊκή, μία επιστολή και με βάση και αυτήν προσπαθώ να σκεφτώ τι είναι το καλύτερο για τις γυναίκες τελικά. Μία πρόταση η οποία θα προσπαθήσει να συμπεριλάβει τα πάντα και τελικά δεν θα περάσει ή μια πιο ρεαλιστική πρόταση, πιο περιορισμένη η οποία έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. γνωρίζετε τη δική μου απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα. Έχω αυτή την νοοτροπία του Λουξεμβούργου. Προσπαθώ δηλαδή τα πράγματα να λειτουργούν. Ας δούμε λοιπόν ποια πρόοδο μπορούμε να επιτύχουμε σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ε, με χαρά μου άκουσα πως σε σχέση με τις ε, κατευθυντές γραμμές ε, για την απασχόληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δίνει περισσότερη έμφαση στον ρόλο των γυναικών. Ε, όπως ε, θα θυμόσαστε, η Επιτροπή είχε αρχικά πει πως πολλά ζητήματα αναφέρονται σιωπηρά. Αλλά αντιλαμβανόμαστε γιατί το Κοινοβούλιο θέλει να κάνει εδώ αλλαγέ. Σε, σε ό,τι αφορά τι ε, συντάξει, εγώ α, στο ε, Green Paper της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχα ε, λάβει πολύ εμφαντικά σε ό,τι αφορά δηλαδή το ρόλο των γυναικών όχι ε, μόνο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και τη φτώχεια. Και νομίζω πως αυτό πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε. Εάν έχουμε δηλαδή ε, μερικές ματιές συντάξεις και τελικά οι γυναίκες χρειάζεται να συνταξιδοτηθούν νωρίτερα, ε, βλέπουμε ε, συχνά να κινδυνεύουν από Άρα βλέπετε ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα και γι' αυτό το Green Paper της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει κάτι τέτοιο. Είδα συχνά αναφορές στον τύπο ότι έχει προτείνει, έχει αποφασίσει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, το μόνο που κάνουμε είναι να αναφέρουμε κάποιες ιδέες ως τροφή για σκέψη για να δούμε τι θα κάνουμε από τότε στο εξή. Πάντως, ε, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πραγματικά εδώ να τοποθετηθεί κατηγορηματικά η Επιτροπή Θέμα σε ό,τι αφορά το ρόλο των γυναικών. Ε, ναι, σε ό,τι αφορά την ε, απασχόληση των ε, γυναικών σε υψηλά αξιώματα. Θεωρώ, εγώ τουλάχιστον ακολουθώ αυτή την ε, πρακτική. Ε, σε ό,τι αφορά το ερώτημα της κυρίας Μπάουρ, νομίζω πως το απάντησα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την ε, μισολογική διαφορά, εδώ χρειαζόμαστε διαφάνεια. Χρειαζόμαστε να λάβουμε ε, μέτρα διαφάνειας και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. σε ό,τι αφορά τους στόχους της Βαρτιλώνας, πραγματικά είναι ντροπή. Είναι κρίμα να έχουμε ε, έτσι, τέτοιους στόχους ε, μη δεσμευτικούς και ούτω καθεξή. Ε, τίποτα δεν συμβαίνει σε τέτοια περίπτωση. Εντάξει, ας μην υπερβάλλω, κάποια βήματα έγιναν σε κάποια κρατημέλη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι τους οποίους είχαμε ζητήσει. Θα πρέπει λοιπόν να επανενεργοποιήσουμε προπονητικά του στόχους αυτούς και να θέσουμε τα κρατημέλη νόμιμα των ταξινών του. Η πρόεδρος θέλει να συντομεύω λίγο. Όχι, εντάξει λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, σας πόσχομαι να συντομεύσω λίγο. Κυρία Παρβάνομα, αναφέρθηκε στη δημογραφική κρίση. Πράγματι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο ζήτημα, αλλά βρίσκεται ενώπιον μας και βλέπουμε προς τα που εξελίσσεται. Και αυτό το λέω γιατί μερικές ε, φορές ε, εργαζόμαστε με βάση το παρελθόν. Ε, δηλαδή βλέπουμε ότι τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν σύντομα και θα πρέπει να έχουμε τις απαντήσεις εκ των προτέρων. Όχι να περιμένουμε να συμβεί το πρόβλημα και μετά να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την έρευνα σε σχέση με τα συστήματα πυλών, έχουμε γι' αυτό το λόγο και το Ινστιτούτο. Και γι' αυτό σας λέω ότι μερικές φορές χρειαζόμαστε χρόνο για τις προτάσεις μας, γιατί χρειαζόμαστε ε, συγκεκριμένα δεδομένα. Ε, συχνά δεν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχουν κάποιες ε, υποθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να, έχουμε, να βασίζουμε νομικές προτάσεις πάνω σε υποθέσεις ε, και γι' αυτό ελπίζουμε πως το Ινστιτούτο θα αναλάβει το συντομότερο δυνατό τις αρμοδιότητες του και θα μπορεί να μας παρέχει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ε, απέναντι στην κυρία ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των διαζυγίων. Βλέπετε πως όταν γίνεται μια σοβαρή πρόταση, ακόμα και όταν είναι πρωτότυπη, γιατί μιλούσαμε για την πρώτη ενισχυμένη συνεργασία, καταφέραμε να έχουμε μια πραγματικά ιδιαίτερη επιτυχία γιατί υποστηρίχθηκε και πολύ από την πλευρά του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο συμφώνησε πολύ γρήγορα. Ε, νομίζω πως ε, απάντησα ήδη στο ζήτημα της εντολής ε, για μεταπροστασία σε ό,τι αφορά τώρα τον ακροτηριασμό των γενικών οργάνων των γυναικών δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το καταστήσουμε αυτή την πράξη ένα έγκλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να μην πέσουμε δηλαδή στην παγίδα του να είναι ε, να διώκεται ποινικά το συγκεκριμένο τη συγκεκριμένη πράξη στο ένα κράτο μέλο και όχι στο άλλο. Να υπάρχει λοιπόν ένα κοινό ορισμό αυτού του εγκλήματο. και ε, θα προσπαθήσω να κινηθώ προς ε, αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ποινικό ορισμό ως έγκλημα αυτής της πράξης. Και σας λέω ότι θα προσπαθήσω και δεν σας λέω ότι θα το κάνω γιατί ε, βρισκόμαστε εδώ πάλι σε έναν καινούριο τομέα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον χώρο του ποινικού δικαίου, ώστε να μην υπάρξει αντίδραση από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί αν ε, γίνει κάτι τέτοιο θα, θα είναι αρνητική η αντίδρασή του. Ε, θα πρέπει λοιπόν και εσεί να ε, μιλήσετε με τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί θα χρειαστούμε την υποστήριξή του σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επιτροπέ, συνεχίζουμε με τις εγγεγραμμένες αγορήτριες και παρακαλώ και πάλι όλες να είναι σύντομες γιατί ο κατάλογος έχει μεγαλώσει κι άλλο. Η κυρία Τόμσον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ανταλλαγή απόψεων που την θεωρώ ιδιαίτερα καρποφόρα για μας εδώ τις Ευρωβουλευτές. Παρακολούθησα τα όσα είπατε για τον χάρτη των δικαιωμάτων γυναικών και το mainstreaming σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα, διότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια στατική για μια πράσινη οικονομία. 8% 80% στην πράσινη οικονομία είναι σε κατοχή ανδρική. Και θα δημιουργηθούν 10 εκατομμύρια νέες εργασίες, νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται η στρατηγική του 2020 κτλ. Από τώρα μέχρι το 2020 λοιπόν. Δεν μιλούν όμως ποτέ για την ανάγκη να αποκτήσουν οι γυναίκες τα προσόντα ώστε να καταλάβουν τέτοιες θέσεις εργασίας. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και την αγορά εργασίας και την οικονομική ανεξαρτησία. Λέμε για το 2020 75% συμμετοχή στην αγορά εργασία των γυναικών. Εγώ νομίζω ότι θα είναι αμοιβαία υποφελή κατάσταση αυτή διότι αφενό θα ενισχυθεί η οικονομική ανεξαρτησία και από την άλλη μεριά και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε συνεχώ. Δηλαδή τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πώ ανταγωνίζεται η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, είμαστε πιο πλούσιοι επομένω και επομένω εξασφαλίζουμε καλύτερο κράτο πρόνοια. Αυτό λοιπόν το 75% είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμω όλοι και όλε πρέπει να βοηθήσουν στι επιχειρήσει. Οι γυναίκες δεν ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Ποτέ δεν ε, ήταν οι γυναίκες στην πλειοψηφία των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών. Και μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Deutsche Telekom έχουν ήδη 30% ποσοστώσεις στις ε, επιχειρήσεις τους. Και λένε ότι δεν, μπορούμε να είναι, δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές εάν δεν έχουν ε, ε, αυτές τις ρυθμίσεις. Τέλος, όταν μιλούμε για την διαφορά στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών και για, για τις γονικές παροχές ε, πατρότητας και μητρότητας δηλαδή. Υπάρχει διασύνδεση μεταξύ ε, άδεια πατρότητας ή μητρότητας και ε, απόστασης χάσματος των αμοιβών. Μόλις αποκτήσουν οι γυναίκες παιδιά, το χάσμα αυτό μεγαλώνει των αμοιβών. Δεν λαμβάνουμε αρκετά υπόψη το χάσμα αυτό όταν λέμε για να μοιραστούν τα δύο φύλλα την ζωή των οικογενειών και να συμφιλειωθούν. Ήρθε μια γυναίκα εδώ στην Επιτροπή μας, την Οντίλ Καντάν, που είπε ότι από την αρχή η Ευρώπη υπήρξε εκείνη η οποία έκανε τις πρώτες κινήσεις για την ισότητα των φύλων. Τώρα όμως κινδυνεύουμε να πέσουμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, αν συνεχίσουμε να ψηφίζουμε νομοθεσία η οποία να εξυπηρετεί τις, ε, ε, όλες τις ε, χώρες. Σήμερα 17 χώρες μέλη έχουν ε, άδεια πατρότητας, οι υπόλοιπες όχι. Τι γίνεται. fru Thomsen. Eh, nästa talare är fru Morin Chartier. Varsågod. Merci Madame la Présidente. Euh, merci beaucoup Madame la Commissaire d'être euh, avec nous. Euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο που είναι εδώ μαζί μας ε, σε αυτό το μεγάλο ερωτοτάξιο για την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και πραγματικά συνεισφέρεται τα μάλα. Θα ήθελα να θέσω κάποιε πολύ απλές ερωτήσεις, αλλά για τις οποίες χρειαζόμαστε ακριβείς απαντήσεις. Η πρώτη μου ανησυχία είναι ότι έχουμε νομοθεσία για την ισότητα στους μισθούς ε, σε αρκετέ χώρες. Όμως τελικά η νομοθεσία αυτή δεν καταπολεμά αυτές τις αποκλίσεις στις αμοιβέ. Έτσι λοιπόν πώς μπορούμε να πάμε πιο πέρα έτσι ώστε στην πράξη να υπάρχει πραγματική ισότητα μισθολογική. Και αυτό και στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό. Πολύ συχνά οι χώρες ε, που μας περιβάλλουν, οι δικοί μου λόγου χάρη, καταδεικνύουν, δακτυλοδεικνύουν τον ιδιωτικό τομέα, λέγοντας ότι στον ιδιωτικό τομέα έχουμε πολύ μεγαλύτερες αποκλήσεις. Αλλά λυπάμαι που δηλώνω ότι και στο δημόσιο τομέα έχουμε πάρα πολλές ε, καθυστερήσεις και αποκλήσεις μισθολογικές πάρα πολύ σημαντικές και ένα τμήμα αφορά και αυτή την άδεια αλλά όχι μόνο. Κάτι ακόμα Μόλις ε, τοποθετήκατε για το θέμα αυτό και είπατε ότι θα πρέπει να διορίσουμε τις γυναίκες στις θέσεις που τους αξίζει. Ναι, εμείς συμφωνούμε, αλλά πώς μπορούμε να αναλάβουμε κοινή δράση έτσι ώστε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικές σε αυτό το τομέα. Έτσι ώστε οι γυναίκες ε, που έχουν ε, τα ίδια προσόντα και τις ίδιες ικανότητες να έχουν πρόσβαση στις ίδιες θέσεις εργασίας. Και Κάτι ακόμη. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε όταν θα εργαστούμε για την, επί της οδηγίας ε, για το ωράρια εργασίας, γιατί η ευελιξία των ωραρίων αυτών ε, να μπορούσε επίσης ε, να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το οικοδόμημα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χιμένες. και του ακροτηρισμού των γεννητικών οργάνων. Η Κομισιόν έχει κατά νου στο να αναλάβει συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα βάσει αυτών των μελετών. Γιατί πάρα πολλές γυναίκες, νέες μετανάστες στην Ευρώπη βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση. Εμείς ε, μας είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε και με άλλους βουλευτές για να τους πείσουμε. Εγώ θα σας βοηθήσω, δεσμεύομαι να σας βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα να αναφερθώ στην κυρία Ρομέρο που είναι η συγγήτρια για το ένταλμα προστασίας. Εγώ παρακολούθησα αυτή την εντολή προστασίας και την παρακολουθώ ακόμα στη συγγήτρια για κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών αισθάνθηκα την ανάγκη να ακούσω πάρα πολλέ ε, απόψεις και έτσι αντιμετώπισα αυτή την έκθεση γιατί νομίζω ότι το σημαντικό είναι να εφαρμόζεται την νομοθεσία και όπως ξέρουμε χαίρει μεγάλη υποστήριξη σε αυτή η πρωτοβουλία γιατί όλοι συμφωνούμε με το στόχο. Το πρόβλημα που έχουμε θέλουμε όμως είναι πώς θα καταστεί με τον καλύτερο τρόπο αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν για μένα και για όλους είναι πολύ πολύ σημαντικό να δούμε και ποια είναι η δική σας άποψη και η δική σας φόβη σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Μήπως μπούμε σε ένα λαβύρινθο για τα θύματα όπως έχουμε πει σε ορισμένε περιπτώσεις. Όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο εργάζεται επί της πρωτοβουλίας αυτής και άκουσα ότι είπατε ότι θα παρουσιάσετε και άλλες γενικές πρωτοβουλίες για τα θύματα. Μια ευρύτερη πρωτοβουλία για το θέμα και φυσικά εγώ το προσυπογράφω και πιστεύω ότι και έχουμε και μία οδηγία θύματα της τρομοκρατίας. Όμως θέλω να σας πω θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η πρωτοβουλία θα συμπληρώσει τη δική μας ε, για να μην αποτελέσει εμπόδιο. Πάντως ε, πρέπει να συνεργαστούμε Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο για να υπερασπίσουμε τα θύματα γιατί πραγματικά αξίζει στα θύματα εμείς να δράσουμε αποφασιστικά και υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παπαδοπούλου. Ε, welcome to meeting and thank you for your... Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ότι θέλετε να παρουσιάσετε ρεαλιστικές προτάσεις γιατί όταν μιλάμε για στρατηγική για την ισότητα των φύλων εδώ και πολλά χρόνια και εδώ αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Συμβούλιο της Ευρώπης πάντοτε συζητούμε ποια είναι τα εμπόδια για την ε, ισότητα των φύλων αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ε, σημειώσει και πολύ μεγάλη πρόοδο και πρέπει να έχουμε συλλογικούς στόχους, συγκριτικές μελέτες και δείκτες για να κρίνουμε την πρόοδο σε κάθε χώρα. Και επίσης πρέπει να έχουμε και αυστηρά χρονοδιαγράμματα προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτή είναι μια γενική δήλωση. Τώρα θέλω να θέσω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν για την οικογενειακή βία. Είπατε ότι θέλετε να εργαστείτε για ένα καθολικό πακέτο για τα θύματα ε, θέλω περισσότερες λεπτομέρειες και θέλω να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα σε ποιο βαθμό πρόκειται να βασιστείτε στο εφιστάμενο έργο που έχει υλοποιηθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την οικογενειακή βία, γιατί ξέρω ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για το όσα κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε επικαλύψεις. Δεύτερη ερώτηση για τον ακροτηρισμό των γεννητικών οργάνων. Γνωρίζω ότι είναι στις αραβικές χώρες και σε ορισμένες θρησκείες ε, λαμβάνει χώρα αυτό το έγκλημα αυτών των γυναικών, έχουμε και τα εγκλήματα τιμής και επίσης έχουμε και παράνομη ε, απαγωγή Ευρωπαίων γυναικών, γυναικών που έχουν γεννηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, όμως δυστυχώς αυτό συμβαίνει έχουμε τέτοιες απαγωγές και παράνομε και παράνομο περιορισμό. Εγώ έκανα μια μελέτη για αυτό το θέμα στο Μαρόκο. Ε, ε είπατε ότι πρόκειται να διασφαλίσετε ότι υπάρχει πλήρης σεβασμός ε, των υποψηφίων χωρών τη νομοθεσία αυτή. Ξέρω ότι τα εγκλήματα τιμή είναι κάτι που συμβαίνει στην Τουρκία. Θέλω λοιπόν να σα ρωτήσω ποια είναι τα πολιτισματικά μέσα που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσει την Τουρκία για να σταματήσει τη διάπραξη των εγκλημάτων αυτών. Γιατί μιλάμε γι' αυτό, αλλά τίποτα δεν συμβαίνει. Τρίτη ερώτηση. Η δημοσιοποίηση, διαφήμιση. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τις διαφημίσεις ε, και όλοι συμφώνησαν ότι πάρα πολύ συχνά στη διαφημίσεις ε, αναπαράγουν σεξιστικά πρότυπα κατά του γυναικείου σώματος και κατά του ανδρικού σώματος. Και η ερώτησή μου είναι είναι εάν είστε πρόθυμοι να προωθήσετε μία οδηγία με αποτελεσματικά εργαλεία και έναν κώδικα δεντολογίας για να διασφαλίσετε ότι η διαφήμιση είναι υπεύθυνη και ηθική. Γιατί έχουμε πρόβλημα εδώ ε, σε ό,τι αφορά την απεικόνιση των γυναικών. Και τελευταία ερώτηση. Για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Πριν λίγες ημέρες έλαβα μια επιστολή στην οποία με ρωτούσαν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα εσείς Επιτροπός είναι πρόθυμοι, είμαστε πρόθυμοι να διερευνήσουμε εις τα εμπόδια τα οποία διατηρούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τη γυναική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Έχουμε τα θέματα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, έλλειψη συμβουλών, ομάδες υποστήριξης και χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνη στις γυναίκες. Ξέρω ότι στι Ηνωμένες τα δεκαετία του 90 υπήρξε μία μελέτη που οδήγησε στο Women Business Ownership Act εσείς είστε πρόθυμοι να παρουσιάσετε μία οδηγία για το θέμα αυτό και να βοηθήσετε στην άρση αυτών των κολλημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι με είχατε ξεχάσει. Ευχαριστώ την κυρία Ρέντινγκ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση θα είμαι σύντομη γιατί όλα τα θέματα καλύφθηκαν. Τα πρώτα όμως τρία θέματα είναι εξαιρετικά γιατί μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε αυτή την ε, ευκαιρία ισοτήτων που χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, η νομοθεσία είναι καλή αν ε, τεθεί σε εφαρμογή. Και χρειαζόμαστε όμως ε, κάτι που να τον υποστηρίζει. Έχουμε ε, την εμπιστοσύνη, το θέμα της εμπιστοσύνης πρέπει να υπάρχει στις γυναίκες. Σκεφτείτε. Σε μία αίθουσα βλέπουμε, παραδείγματο χάρη, πολλές γραβάτες ε, και κουστούμια και εγώ θα ήθελα να πω αν μια γυναίκα μπει εδώ στην αίθουσα αυτή με κουστούμι και γραβάτα βάζω στοίχημα ότι θα πετύχει αυτό που θέλει γιατί είμαστε γυναίκες δυναμικές και πρέπει να ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση, με την παιδεία έτσι ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα. Σε ένα άρθρο μιας εφημερίδας ε, διάβασα ε, ένα άρθρο ότι οι γυναίκες ε, λαμβάνουν, μάλλον μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών σήμερα είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου από ότι άνδρες. Και αν δούμε το θέμα της οικονομικής ανεξαρτησίας, τότε θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση να έχουμε και γυναική επιχειρηματικότητα. Όπως ε, ξέρετε, πολύ καλή δουλειά έχει γίνει στην Αμερική στο τομέα αυτό και θέλω οι γυναίκες να έχουν την εμπιστοσύνη και να έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να εργαστούν στον ε, τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να εργαστείτε στον τομέα της παιδείας, στην ενδυνάμωση των γυναικών και στο πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις γυναίκες να πετύχουν στον τομέα που έχουν επιλέξει. Ευχαριστώ κυρία Φιγερέιδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Φυσικά, εγώ με ανυπομονησία περιμένω να δω αν μπορούμε να δώσουμε κάποια προώθηση, κάποια όθηση διαρκεί στο χρόνο τα δικαιώματα των γυναικών στη νέα πρόταση που θα μας στείλετε. Και θεωρώ ότι αυτό που μας αναφέρατε μπορεί να είναι σημαντικό. Δηλαδή, στο ότι ζητήσατε από τους υπόλοιπους επιτρόπους να αναλάβουν δεσμεύσεις γιατί τους υπενθυμίσατε, γιατί πρέπει να είναι εγκάρσιο το θέμα της ισότητας και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ λοιπόν Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι έχω κάποια περιέργεια για να δω πώς ε, το αίτημα αυτό θα απαντηθεί από τους συναδέλφους σας. Και στη συνέχεια εδώ μπορούμε να αναλύσουμε και να δούμε σε κάθε τομέα τι γίνεται. Φυσικά αυτό είναι ένα έργο που πρέπει να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, το δεύτερο σχολείο μου έχει να κάνει με το εξής. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ανησυχητική η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όχι μόνο βάσει των στοιχείων που βλέπουμε ότι υπάρχουν επισφαλείς εργασίας για τις γυναίκες, χαμηλή μισθή, ανεργία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και οι ε, στην ε, εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη μητρότητα. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε δύο τεινά που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τις χώρες και τις επιχειρήσεις που σέβονται την νομοθεσία, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα είδος μαύρου βιβλίου εκεί θα καταγγείλουμε λόγου χάρη τις περιπτώσεις αυτές όπου υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την μητρότητα. Βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνονται τέτοιου είδους οι καταγγελίες. Και μάλιστα και στη δική μου χώρα αλλά και σε άλλες χώρες, ορισμένες από αυτές τις καταγγελίες φτάνουν μέχρι και εδώ στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν το Ινστιτούτο για την Ισότητα θα μπορούσε να διερευνήσει αυτή την υπόθεση. Κάνω κάποιες προτάσεις εδώ προς αξιολόγηση ε, ίσως να μπορούμε να τις δούμε στο μέλλον τις ιδέες αυτές. Τώρα, κάτι ακόμα. Αν Δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τις μισθολογικές αποκλήσεις, τις μισθολογικές διακρίσεις σήμερα. Αυτές οι μισθολογικές διακρίσεις είναι περισσότερο έμεσες παρά άμεσες. Δηλαδή, υπάρχει και μια διαφορετική μεθοδολογία. Εγώ γνωρίζω ότι ε, εκπονούνται κάποιες μεθοδολογίες στον τομέα αυτό, οι οποίες ε, ουσιαστικά δίνουν μεγαλύτερη αξία στα επαγγέλματα όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, έτσι ώστε να μπορέσουν ε, να ε, αξιοποιηθούν, μάλλον να ανέλθουν και οι αμοιβέ. Τώρα, μία στρατηγική για την ισότητα θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει το δικό της προϋπολογισμό και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ενίσχυση των κονδυλίων. Στο Progress λόγου χάρη και συγκεκριμένα στους τομείς ε, που απευθύνονται στις γυναίκες αλλά και στην καταπολέμηση της ανέχειας στο θέμα του ευρωπαϊκού ελαχιστού εισοδήματος είναι ένα θέμα που έχει τεθεί επιτάπητος, που έχει ως στόχο να καταπολεμήσει την φτώχεια των γυναικών καταρχήν, γιατί είναι γυναίκες που θίγονται περισσότερο. Εγώ θα ήθελα επίσης να εμπλοκείτε και σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά έχουμε και το θέμα της οδηγίας για τη μητρότητα για την άδεια και για την άδεια Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι θετικές πτυχές και να προσπαθήσουμε να είμαστε φιλόδοξοι Δηλαδή να μην συνεχίσουμε μια πολιτική ε, η οποία θα θεωρεί ότι η μητρότητα είναι άχθος για τις γυναίκες. Όχι. Για να έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεωρήσουμε ότι η μητρότητα ουσιαστικά είναι κάτι προς διεξία και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε θα προσπαθήσω να πω και εγώ δύο λόγια μετά από τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την ισότιμη μεταχείριση, ε, προφανώ πρόκειται για μια πολιτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι επίτροποι από κοινού. Ήδη είπε η επίτροπο Ρέντινγκ ότι η οι επιτρόποι θα υποβάλουν μια πρόταση από κοινού και προφανώ αυτή την πρόταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα ισότιμη μεταχείριση. Είναι σημαντικό αυτό προκειμένου η στρατηγική για την ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών να είναι δυνατόν να εφαρμοστεί παντού και να χαίρει και του ίδιου σεβασμό. Υπάρχουν όμω και άλλα ζητήματα, ζητήματα υγεία για παράδειγμα ε, των γυναικών. Όταν αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα ε, έχουμε να κάνουμε κυρίω με δικαιώματα αναπαραγωγή αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες επιτυχίες σε ό,τι αφορά το, το τομέα της υγείας. Δηλαδή, διάκριση μεταξύ των φίλων σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. θα το λάβετε αυτό υπόψη σας, Επίτροπε, στη δική σας ε, μια ακόμα ερώτηση. Η Επίτροπο Ρέντινγκ μας υποσχέθηκε πως ε, θα ε, υπάρξει μια πρόταση από την πλευρά τη το 2011 ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη βία ει βάρος των γυναικών. Η δική μου ερώτηση είναι, θα καλύψει αυτή η πρόταση τους διάφορους τομείς στους οποίους ε, αφορά αυτή η βία, δηλαδή η βία με τις διαφορετικές μορφές με τις οποίες εκφράζεται. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Σε ό,τι αφορά το τομέα της απασχόλησης, συχνά κάνουμε λόγο για την ανάγκη να ε, αναδείξουμε τις ε, πρακτικές εκείνες οι οποίες ε, έχουν λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο και έχουν αποδείξει την αξία τους. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Επιτροπή να εξετάσει το πώς έχουν τα πράγματα στα διάφορα κράτη-μέλη, να αναλύσει τις πρακτικές που εφαρμόζονται εκεί και να διαπιστώσει εάν με βάση τα μέτρα ε, που ελήφθησαν σε αυτά τα κράτη, αυξήθηκε πράγματι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Και επίσης ε, να εξετάσει η Επιτροπή ε, το πώς έχει το νομικό καθεστώ στα διάφορα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την άδεια μετρότητα. Η κυρία Ζαγούσα έχει το λόγο. Okay. okay. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Επίτροπε, και σας ευχαριστώ και για την απαντήση που δώσατε στην κυρία Μπάουερ για την οδηγία για την αδιαμητρότητα. Ξέρω ότι είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πρόβλημα. Ήθελα να θέσω μια πρόσθετη ερώτηση αλλά βλέπω τώρα ότι η κυρία Στρέλα δεν είναι εδώ ως συγκεντρία. Έτσι λοιπόν, δεδομένου και του χρόνου, θα έλεγα ότι προτιμώ να αναβάλω την ερώτησή μου για κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ. Κώστα. Ε, gentile commissaria, Ευχαριστώ. Θέλω να θέσω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι εξή Εσείς ανακοινώσατε αυτή τη σημαντική βούληση να αναθεωρήσετε πιο οριζόντιο τρόπο την πολιτική της διακυβέρνησης και νομίζω ότι και η στρατηγική για την Ευρώπη το 2020 θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μια πιο επιχειρησιακή εποπτεία, παρακολούθηση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον ε, νέο προγραμματισμό για τα Ευρωπαϊκά Διαθροτικά Ταμεία. Εγώ έχοντας ε, μια τέτοια εμπειρία θεωρώ ότι έχοντας ε, θέσει το mainstreaming ε, μόνο και και έχοντας ε, αφαιρέσει ε, στοχευμένες συγκεκριμένε δράσεις για τις γυναίκες, εγώ θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ευνοήσει μια συνεχή προσοχή για τον αντίκτυπο που έχουν τα διαφορετικά ταμεία στις γυναίκες. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό στο μέλλον. Κάτι ακόμη με ενδιαφέρει η αξιολόγηση αντικτύπου της οδηγίας ε, που ελπίζω σύντομα να μπορέσει να εγκριθεί για τις άδειες μητρότητας. Αλλά αναρωτιέμαι, πέρα από το θέμα της ε, εισαγωγής της άδειας πατρότητας που δεν είναι μόνο συμβολικό, θα ήθελα ε, να μην ακολουθήσουμε μία προσέγγιση εδώ μόνο μαθηματικού χαρακτήρα, γιατί δεν θα ήθελα το μήνυμα που θα δοθεί στις γυναίκες της Ευρώπης να είναι ότι η μητρότητα, ε, η προστασία της μητρότητας ή ε, η φροντίδα κοστίζει πάρα πολύ και ότι αντίθετα οι γυναίκες ε, θα πρέπει να είναι ισότιμες μόνο σε ό,τι αφορά το ότι πρέπει να εργάζονται περισσότερα χρόνια. Εμείς ε, θεωρούμε ότι εντάξει αυτό έχει ένα ε, θετικό, αλλά όχι για όλες τις γυναίκες, όμως ε, θα πρέπει το, η επιμήκυνση της ζωής, της επαγγελματικής ζωής των γυναικών να συνοδεύεται και από άλλα μέτρα για να μπορούν και οι γυναίκες να φτάσουν σε ένα σημείο να συνταξιδοτούνται. Θα ήθελα να αναφερθώ επίση στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η φτώχεια θίγει κυρίως στι γυναίκες και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Αναρωτιέμαι μήπως θα υπάρχει μία πρωτοβουλία που θα αναλυφθεί, ίσως να μην γνωρίζω επαρκώς, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, θα υπάρξει ανάληψη κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να καταπολεμήσετε τη φτώχεια των γυναικών και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό, γιατί εγώ θεωρώ ότι κυρίως οι γυναίκες θίγονται στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος το πάλι σε εσάς, ε, κύριε Επίτροπε. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Και όσο γίνεται βέβαια σε περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Για να απαντήσω καταρχήν ε, ε, στο ερώτημά σας σε ό,τι αφορά το πού βρισκόμαστε σε σχέση με το παράτημα της ε, στρατηγικής. Ε, είναι πολύ σημαντικό από πολιτική άποψη σε αυτό, γιατί δείχνει το ρόλο που αναλαμβάνουν οι συνάδελφοί μου σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των, της πολιτικής για την ισότητα μεταχείριση σε ό,τι αφορά τις, τα διάφορα παιδεία. Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευση, ε, το μέρα αρμοδιότητας ε, τη κυρία Βασιλείου ή το τομέα αρμοδιότητας του κ. Ότιγκερ ή για παράδειγμα το ε, Επίτροπο Απασχόληση στη Ρουάντα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε στου συναδέλφους επιτρόπους αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να το πράξουμε με έναν επικοδομητικό τρόπο γιατί μερικές φορές η διοίκηση θεωρεί πως, ε, πως ε, τα ε, ζητήματα, όλα τα ζητήματα που αφορούν την ό,τι μεταχείριζε μεταξύ των δύο φίλων είναι αρμοδιότητα δική μου και κανένα άλλου. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν ότι είναι, εντάσσεται αυτή η πτυχή και στη δική τους πολιτική και θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να τους βοηθήσει να το αντιληφθούν αυτό, του συναδέλφου μου δηλαδή σε ό,τι αφορά την ε, άδεια μητρότητας και την ε, διαφορά στους ε, μισθούς, είναι σαφές πως αν κανείς λείπει συχνά από την δουλειά, όχι μόνο θα υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά δηλαδή χαμηλότερο εισόδημα, αλλά θα υπάρξει και πρόβλημα σε ό,τι αφορά την σύνταξη τη χαμηλότερη σύνταξη. Και βέβαια οι ε, στόχοι της ε, Βαρκελόνη έχουν εδώ να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή να ασκήσουμε πιέσεις στα κράτη-μέλη, ώστε να συμμορφωθούν με τις ε, υποσχέσεις τους. σε ό,τι αφορά α, αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ισότητας σε ό,τι αφορά τους μισθούς, είναι ε, παλιό θέμα. Ε, περιλαμβανόταν ήδη στις δικές της Και οι οδηγίες ε, που προήρθαν, προήρθαν από τότε, από εκείνες τις συνθήκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βασίσουμε σε αντίστοιχε διατάξεις που έχουν πλέον καταστεί εργατικό δικαίωμα στα, στα κράτη-μέλη. Και αν βέβαια διαπιστώσουμε πως υπάρχουν ε, ε, παραβάσεις από την πλευρά των κρατών μελών, δεν θα διστάσω να εκινήσω διαδικασίες κατά παραβάση. Ε, θα ήθελα επίσης οι γυναίκες να ενεργοποιηθούν, να το πούμε, να δραστηριοποιηθούν λίγο από μόνες τους, εθελοντικά, να αξιώσουν αυτά τα πράγματα, να μην περιμένουν να κάθονται στη γωνία και να περιμένουν να τις επιλέξουν. Να είναι δραστήρες από μόνες τους για να δείξουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ό,τι χρειάζεται. Η διάσκεψη τώρα του Νοεμβρίου διοργανώνεται ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει και η Προεδρία του Συμβουλίου. Τα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη θα αναλυθούν προφανώς στο πλαίσιο της διάσκεψης και θα υπάρξει προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων βίας. για το συνολικό πακέτο μέτρων το οποίο θα σας παρουσιάσω του χρόνου. Η ευρεία διαδικασία ε, διαβούλευση σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα ξεκινήσει από αύριο. Σε ό,τι αφορά την θέση και στην αγορά ε, προφανώ θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά εδώ τι εξελίξει και θα πρέπει να δώσω στον τις τι ε, σχετικέ οδηγίε, ώστε να μπορέσει να συμπεριλάβει αυτή την πτυχή ε, στο δικό του έργο. Σε ό,τι αφορά την για τη βία, τη βία εις των ε, γυναικών, ε, την, ε, τον ακροτηρισμό των γεννητικών οργάνων. Ναι, θα ενσωματώσουμε τις εργασίες που έχει κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ και θα ήθελα και η Ένωση των Μεσογειακών Χωρών να εμπλακεί περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Όταν θα υπάρχει διάλογος μεταξύ ορίων χωρών Μεσογείου και Νοτιών χωρών να θίγεται και αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποψηφίων χωρών, ε, προφανώς ε, καλούνται υποχρεωμένε αυτές οι χώρες να ε, ανταποκριθούν πλήρω στι υποχρεώσει που προβλέπονται και η ε, φόνη τιμής και αντίστοιχη γάμοι όπω γίνονται καταναγκαστικοί αποτελούν ζητήματα εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ε, γενικότερης ε, ε, ενσωμάτωσης αυτών των ε, ζητημάτων στο κοινωτικό κεκτημένο επιλαμβάνεται αυτών των ζητημάτων. Οι συνεργάτες μου στην διάσκεψη που έγινε τον Μάιο αναφέρθηκαν εκτενώς σε αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά σε σχέση με την υγεία. Γνωρίζετε πως έχουμε την έκθεση για την υγεία του 2010 και ο ε, θέλει να προωθήσει περαιτέρω αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τη γυναική επιχειρηματικότητα υπάρχει μία πρωτοβουλία την οποία θα αναλάβουμε, όχι μέσα στις επόμενες εβδομάδες ίσως, αλλά η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας γιατί πραγματικά θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε περισσότερο τις γυναίκες να προχωρήσουν μπροστά και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Και εδώ να υπογραμμίσω πως οι μικροπιστώσεις, τα micro-credits ε, ε, είναι πραγματικά θεμελιώδους σημασία και το έχουν αποδείξει αυτό στην, στις χώρες του τρίτου κόσμου. Οπότε γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και εμείς εδώ Το πρόβλημα δηλαδή που αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκε είναι ότι δεν ε, υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη απέναντί τους, ε, δεν έχουν δηλαδή την κατάλληλη αξιοπιστία για να λάβουν ένα δάνειο. Αντίθετα όταν ε, ο υποψήφιο για το δάνειο είναι άντρα, έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Προφανώ η ε, φροντίδα των παιδιών σχετίζεται άμεσα με την συμμετοχή του στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Βρήκα την συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Άλλωστε πολλά μέλη της Επιτροπής μας συμμετέσχαν στη συζήτηση και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον για την συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την έλευσή σας σήμερα εδώ, για την δέσμευσή σας ως Επιτρόπου σε θέματα ισότητας των φύλων και θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία να σας εκφράσω την ευχή μάλλον, να περάσετε καλές και στι θερινές διακοπές. Σας ευχαριστούμε και πάλι. you before. Έχουμε ένα θέμα ακόμη. Έχουμε ακόμα ένα θέμα ε, στην ημερήσια διαταξή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν την συνεδρίασή μας. Το επόμενο θέμα είναι η θέση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο του προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Τμήμα 3, Επιτροπή. Υπενθυμίζω ότι τον Μάιο η Επιτροπή μας ενέκρινε γνωμοδότηση για, την, για τον προπολογισμό του 2011, γνωμοδότηση την οποία διαβίβασε στην Επιτροπή Προπολογισμών και η οποία εν τέλει βρήκε τη θέση της στο ψήφισμα της 15ης Έκτου. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και εντολή για τον τριμερή διάλογο του επόμενου έτους. Η διαδικασία προχωρεί. Έχουμε τώρα μια τροποποιημένη πρόταση και τα αριθμητικά στοιχεία έχουν ε, αλλάξει. Η κυρία Γκαρσία Πέρες δυστυχώς είναι απούσα, που είναι η συντάκτη της γνωμοδότησης. Η κυρία Τόμσον όμως είχε αναλάβει να την εκπροσωπήσει και θα την παρακαλέσω να λάβει το λόγο. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες για την αποκατάσταση των ε, αριθμών, των αριθμητικών στοιχείων. Δεν δεχόμαστε δηλαδή τις περικοπές για τις πολιτικές ε, ισότητας ε, των φύλων. Δεν θα πρέπει να περικοπούν τα ποσά αυτά. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες που συνδέονται με το πρόγραμμα πρόοδου. Και θα πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν η μείωση του προπολογισμού οφείλεται στη δημιουργία νέου μηχανισμού που λέγονται μικροπιστώσεις υπέρ των νέων στην Ευρώπη. Και αν αυτά χρηματοδοτούνται ε, αποκλειστικά από τα ε, προγράμματα ισότητας ή και από άλλα. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν τα ποσά του προϋπολογισμού για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του, του προγράμματος Δάφνη και, τον, ε, και του Ινστιτούτου που ασχολείται με την ισότητα των φύλων. Έχουμε και 7 pilot projects που προτάθηκαν από διάφορες συναδέλφους, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα περισσότερα από τα project αυτά βρίσκονται ήδη στην φάση της εξέλιξης. Ένα είναι μια επέκταση ενός ε, ισχύοντος προγράμματος για την ε, αντιμετώπιση των αβέβαιων θέσεων εργασίας και των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές. Άλλα προγράμματα έχουν σχέση με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ε, για την αναγνώριση της εργασίας ε, των προσώπων που προσφέρουν φροντίδα σε εξαρτώμενα πρόσωπα της οικογένειας και που είναι ιδίω γυναίκες, να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τα pilot project οι συνάδελφοι, γιατί δεν θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε όλα, δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να επιτύχουμε την έγκριση όλων και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένα. Έχουμε και άλλα όπως η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τις ε, ηλικιωμένες γυναίκες, για την ε, επανένταξη γυναικών που υπήρξαν θύματα βίας στην αγορά εργασίας και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδη συγγητρία για το ΕΛΚΑ για τον προπολογισμό του 2011 και ζήτησα το λόγο για να κάνω και ένα σχόλιο για τον ευρωβουλευτικό της Εγώ καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένη για τα κονδύλια που έχουν εργοποιηθεί για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Πρόκειται για σημαντικά κονδύλια που μπορούν να βοηθήσουν να συμβάλλουν στην πρόθεση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, γιατί μπορούμε να θυμηθούμε ότι πέρσι υπήρξαν και ορισμένα προβλήματα πρόσληψης ε, στο Ινστιτούτο και έτσι εγώ νομίζω λοιπόν ότι τώρα τα κονδύλια που έχουν δεσμευτεί θα έχουν ε, θετική θετικό αντίκτυπο για τις δραστηριότητες του ίδιου του Ινστιτούτου. Όμως, ε, από την άλλη, λυπούμε για τις ε, μειώσεις που έχουν γίνει. Μιλάμε, ε, το εδώ έχουμε μείωση των κονδυλίων στο πρόγραμμα Δάφνη για την καταπολέμηση της βίας. Εγώ νομίζω ότι αυτή η μείωση των κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί, που ζήτησε καταρχήν η Κομισιόν και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από την Κορεπέρ σε πολύ, ε, στο πολύ εγγύς μπορεί να μας οδηγήσει στο να έχουμε μη επαρκή αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών αλλά και των πλέον ευαλώτων ατόμων όπως τα παιδιά και επίσης θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο και στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Έτσι λοιπόν Λυπούμε γι' αυτό, όπως λυπούμε και για τη μείωση των κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί για το πρόγραμμα Progress και συγκεκριμένα αναφέρομαι στις γραμμές προϋπολογισμού για την ποικιλομορφία, για τη διαφορετικότητα και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την ισότητα των φύλων. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι μαθηματικές ε, είναι σήμερα ενεργές στο εσωτερικό της ε, ίδιας της Ένωσης και της κοινωνίας μας και έτσι λοιπόν ε, αυτή η μείωση στον προπολογισμό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε αυτούς τους τομείς. Ε, έτσι λοιπόν δεν υποστηρίζονται οι δραστηριότητε των δύο των προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν εδώ συμφωνώ με την εισηγήτρια και ξαναπροτείνουμε να επανέλθουμε στα ποσά που είχαμε το 2010. Και επειδή μιλήσατε και για πιλωτικά προγράμματα, εδώ δική μας Επιτροπή, αλλά και εγώ ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η, Επιτροπή για τις ίσες ευκαιρίες γιατί ήταν ε, πάρα πολύ ε, λίγα τα πιλωτικά προγράμματα. Έτσι λοιπόν θέλω να απευθύνω έκκληση στις συναδέλφους να επαναπροσδιορίσουν αυτά τα προγράμματα και να φερθούν πιο συγκεκριμένα σε αυτά και να παρουσιάσουν τροπολογίες ε, για τον προπολογισμό. Νομίζω ότι μέχρι τις 21 αυτού του μήνα είναι η προθεσμία. Έτσι λοιπόν θέλω να απευθύνω αυτή την έκκληση στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ματέρα. Κύριε Φιγκερέιντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ Έχω πάρα πολλέ ανησυχίε ε, εδώ. Αναφέρθηκαν βέβαια πολλά από αυτά που θέλω να πω. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη θέση ε, της Κομισιόν του Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή σε σχέση με το πρόγραμμα Progress. Γιατί, εγώ θυμάμαι ότι 11 χρόνια πριν, όταν το πρόγραμμα Progress αντικατέστησε 5 άλλα προγράμματα, και ε, οι συνάδελφοι που ήταν εδώ και συμμετείχαν σε εκείνη τη συζήτηση γνωρίζουν πόσο πολύ συζητήθηκε αυτό το θέμα. Πάντοτε αυτό έγινε με την υπόσχεση ότι οι τομεί τη ισότητα. δεν μιλάμε για την ισότητα των φίλων, δεν μιλάμε για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Θα λαμβάνονταν πάντοτε υπόψη και θα λάμβαναν τη σωστή χρηματοδότηση. Και τώρα βλέπουμε το αντίθετο. Βλέπουμε ότι υπάρχει προοδευτική υποτίμηση αυτών των τομέων από τη σκοπιά του προπολογισμού. Ενώ έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα τα επαναλάβω τώρα εδώ, γιατί μόλις τώρα το συζητήσαμε αυτό το θέμα με την Επίτροπο. Έτσι λοιπόν πρέπει εμείς εδώ να επιστήσουμε την προσοχή μας ε, στην ενίσχυση αυτών των κονδύλιων. Αν ήδη το 2010 το κονδύλι ήταν χαμηλό, τότε είναι δυστυχές αυτό που συμβαίνει φέτος. Πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να επιμείνουμε σε μια μεγάλη ενίσχυση αυτών των κονδυλίων. Δεν ξέρω διαδικαστικά πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε να μας ενημερώσει η γραμματεία. Εμείς πάντως από τη δική μας πλευρά θέλουμε να συνεισφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να υπάρχει ουσιαστική αύξηση. Επίσης, πρέπει να, λάβουμε, να έχουμε κατά νου ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει φέτος με το τι συνέβαινε πέρσι, εμείς θέλουμε και το επόμενο έτος το σύστημα να λειτουργεί πλήρως. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα κονδύλια που έχουμε δει δεν διασφαλίζουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι διαβιές σαν το είδωρ. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή την αύξηση στα κονδύλια. Και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε μια χρονική στιγμή που εμεί προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των γυναικών, από το ταμείο αυτό ίσω θα μπορούσαν να προέλθουν κονδύλια για τον τομέα αυτό. Επομένω δεν καταλαβαίνουμε καθόλου τι γίνεται. Γιατί το Συμβούλιο ουσιαστικά προτείνει τη μείωση των κονδυλίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ακατανόητο και κυρίως ό,τι αφορά τις πληρωμές, τις πιστώσεις πληρωμών. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά σχέδια και το πρόγραμμα Δάφνη. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε και εδώ να επιμείνουμε έτσι ώστε τα ζητήματα της ισότητας που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις γραμμές προϋπολογισμού να ενισχυθούν. λίγα πιλωτικά σχέδια ούτως ή άλλως είχαμε παρουσιάσει στον τομέα της ισότητας. Και θα πρέπει λοιπόν να τα περισπίσουμε όλα αυτά. Και ενώπιον της Κομισιόν και του Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή. αλλά και στην Επιτροπή Προπολογισμών εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει οι συνάδελφοι μας να ευαισθητοποιηθούν για αυτούς τους τομείς τους οποίους συζητούμε εδώ. Χρειάζεται να υποστηρίξουμε την εισηγήτρια στην Επιτροπή Προπολογισμού. Θα πρέπει η συνάδελφο να ευαισθητοποιήσει και του υπόλοιπου συναδέλφου στην Επιτροπή Προπολογισμού. Ίσως βέβαια και εμείς μπορούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη δουλειά στις πολιτικές μας ομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση και το περιεχόμενό της. Ε, ουσιαστικά εδώ προσπαθούμε να διορθώσουμε το, τι, το κακό που προβλέπεται. Όμως ορισμένα σημαντικά κεφάλαια σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Δάφνη, Progress, ε, η Επιτροπή έχει προτείνει χαμηλότερα ποσά για το 2010. Έτσι λοιπόν, δεν βλέπουμε εδώ καμία αύξηση και μάλιστα πέρα από την πρόταση της Κομισιόν μας έδωσε και αυτό το μήνυμα το Συμβούλιο και μάλιστα, κοιτάξτε, έχουμε και το έτος καταπολέμησης της στόχιας ε, και τώρα εδώ, ενώ έχουμε αυτό το έτος, ερχόμαστε να μειώσουμε τα κονδύλια για το Progress. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργούσε, όμως ε, είχαμε πάρα πολύ δύσκολο έργο να συντονίσουμε τα διάφορα προγράμματα, όπως το Equal και τα υπόλοιπα. Εδώ Εύχομαι το φθινόπωρο να εγκριθεί οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά ε, εδώ βλέπουμε να υπάρχει μείωση των κονδυλίων στο πρόγραμμα Δάφνη και είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα ε, της Ευρώπης ε, και μάλιστα βλέπουμε εδώ ότι έχει υπάρξει και αύξηση αυτών των εγκλημάτων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και αυτό το ευρωπαϊκό έτος και από την άλλη βλέπουμε να μειώνονται τα κονδύλια. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σε μια αντίφαση, αντίφαση της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναφέρω και κάτι ακόμα, να υπενθυμίσω κάτι που αναφέρει η κυρία Φεγκερέιντο. Ας θυμηθούμε και τη δέσμευση που αναλήφθηκε γιατί μαζί με το progress, το οποίο δεν πρέπει να αφηγεί, όσο οντότητα ίσως να, υπάρχει και, να υπάρχουν και κάποιοι πόροι ε, για την μικροχρηματοδότηση. Δεν ξέρω αν είχαμε σύσταση, αλλά είχαμε μία νέα γραμμή που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο για να προωθήσουμε τη μικροπίστοση, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Ρέντινγκ προηγουμένως. Έτσι λοιπόν θέλουμε να δούμε τι ακριβώς προβλέπεται και στον προϋπολογισμό. Ίσως εγώ να μην το είδα αυτό, αλλά αν έχουμε αυτή την μικροπιστώση, αυτό δεν ευνοήσει πάρα πολύ τις γυναίκες. Δεν βρίσκω αυτό το κεφάλαιο που για μας ήταν στρατηγική σημασία. Ίσως λοιπόν για το θέμα αυτό θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή πρωτοβουλία από τη δική μας Επιτροπή. Να μην περιοριστούμε λοιπόν στο να ζητήσουμε αποκατάσταση των κονδυλίων αλλά Ίσως θέλω να προτείνω εδώ να έχουμε και μια επιστολή της Προέδρου προς ε, όλους τους επικεφαλείς ε, των ομάδων αλλά και προς την Επίτροπο Ρέντινγκ γιατί μόλις εμείς τώρα είχαμε μια κρόση με την Επίτροπο Ρέντινγκ και ίσως θα ήταν καλό να τις ζητήσουμε και να μας βοηθήσει σε αυτή τη μάχη για να έχουμε έναν ε, μεγαλύτερο προπολογισμό, ο οποίο ε, να μην ε, έρχεται σε αντίφαση με όλα αυτά τα οποία σα ανέφερα μόλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Το λόγο θα ήθελα να δώσω τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, με συγχωρείτε κυρία Πάουερ πρώτα. συγγνώμη που διακόπτω. θα ήθελα να σας θυμίσω ότι την τελευταία φορά που συζητήσαμε θέματα προϋπολογισμού θυμούμε ότι έχουμε ένα πενταετές πλαίσιο για το πρόγραμμα Δάφνη για την χρηματοδότηση της προστασίας των θυμάτων και της σωματεμπορίας. Εγώ θέλω να ζητήσω να μην αυξηθούν οι περικοπές που θα γίνουν φέτος. Το είχα ζητήσει αυτό μάλλον, αλλά δεν είναι δεκτή η αίτησή μου. Και η παρούσα επιτροπή αύξησε τα ποσά που θα αποσυρθούν φέτος. Βέβαια το πλαίσιο έχει θεσπιστεί εδώ και πολύ καιρό. Σας θυμίζω πάντως ότι προσπαθήσαμε να βρούμε άλλες πηγές για τη χρηματοδότηση των, ε, της προστασίας των θυμάτων, για παράδειγμα με την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των δραστών και τα χρήματα αυτά να πάνε υπέρ της προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι είχαμε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουμε 100 εκατομμύρια από το Progress Budget για τις μικροπιστώσεις. Και αυτό ψηφίστηκε και εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάουερ. Από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τις ερωτήσεις. Έρχομαι στην πρώτη τελευταία παρέμβαση. Υπάρχει πράγματι στο προσχέδιο προϋπολογισμού κονδύλιο για το μηχανισμό μικροπιστώσεων, περίπου 25 εκατομμυρίων. Δεν το έχουμε λησμονήσει αυτό, ούτε το περιέκοψε το Συμβούλιο. Επανέρχομαι στην πρώτη σας ερώτηση για τις περικοπές στο Progress. Το ιστορικό για να τροφοδοτήσουμε τον μηχανισμό αυτό των μικροπιστώσεων είχαμε συμφωνήσει να διατεθούν 60 ε, τελικά εκατομμύρια από το Progress Budget για τις μικροπιστώσεις 40 εκατομμύρια από το περιθώριο και μια μονομερή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το περιεχόμενο ότι στην διάρκεια υποβολής προτάσεων του προϋπολογισμού θα γινόταν κάθε τι το δυνατό για να ε, διατεθούν 20 εκατομμύρια από το περιθώριο μέχρι το 2013 για να επαναποκατασταθούν εν μέρη τουλάχιστον τα ποσά του Progress. Αυτά ιστορικά. Δεύτερο, δεν υπήρξε άνηση μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων τμήματων του Progress. Υπήρξε μια αναλογική μείωση καθενός τμήματος με τρόπο πάντως που σεβόταν την ανακατανομή που είχε γίνει με την απόφαση. Δεν έπασχαν περισσότερο δηλαδή τα ε, ε, ενδιαφέρουν για την ισότητα των φίλων κλπ. από τα υπόλοιπα. Βλέπω πράγματι που προτείνεται, ότι προτείνεται να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τις υποχρεώσεις λίγο περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Εν τέλει γιατί όχι. Ξέρετε πάντως υπάρχει διαφορά μεταξύ πιστώσεων υποχρεώσεων και πληρωμών το Συμβούλιο μείωσε σημαντικά τις πιστώσεις πληρωμών σε όλα τα κονδύλια και του Progress. Πάντως, στην πρότασή σας, εσείς προτείνατε να επαναποκατασταθούν οι πιστώσεις πληρωμών στο επίπεδο του σχεδίου. Σε ό,τι αφορά τα pilot projects, Όντως ένας αριθμός από αυτά είχαν προταθεί. Θα είδατε την ανάλυση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω να χρειάζεται να λεχθεί ότι ορισμένα έχουν γίνει δεχτά, αλλά όχι. Έχει γίνει μια σε βάθος ανάλυση και ένας αριθμός προτάσεων προτινόμενων project pilot, ε, pilot projects μάλλον, καλύπτονται ήδη από ε, υφιστάμενα προγράμματα και ιδίως το Progress. Σε αυτή τη βάση λοιπόν ορισμένα project μπήκαν σε κατηγορία C. Τα α και β μπορούν να υλοποιηθούν με κάποια τροποποίηση, ενώ τα C είναι αυτά τα οποία καλύπτονται ήδη από άλλα. Δύο λόγια για τις μικροπιστώσεις. Δεν μειώσαμε το progress για να κάνουμε κάτι το απόλυτα ξένο στον προβληματισμό της ε, ισότητας των φύλων, γιατί οι μικροπιστώσεις, όπως ε, είπε κάποια συναδελφό σας, είναι ένας μηχανισμός χρηματοδοτικός που μπορεί ε, να ενισχύσει γυναίκες για να ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα και εδώ είναι και η διασύνδεση με το Κοινωνικό Ταμείο όπου στα πλαίσια της υλοποίησης αυτού του μηχανισμού μικροπιστώσεων θα έρθουν δράσεις της Κομισιόν για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αρχών διαχείρισης του Κοινωνικού Ταμείου, του Κοινωνικού Ταμείου για να προσφύγουν στις δυνατότητες που δίνει ο μηχανισμός μικροπιστώσεων. Τώρα, ε, ευχαριστώ την προσοχή σε ένα θέμα όπου το Συμβούλιο περιέκοψε σημαντικά στο κονδύλιο δηλαδή, είπα για το πρώην ταξιακό εργαλείο. Γίνεται μια πρόταση περικοπών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και για έναν αριθμό των προβλεπόμενων δράσεων που θα ενίσχυαν τις προσπάθειες που γίνονται για την ισότητα των φίλων στις ε, ε, υποψήφιες χώρες και που ίσως έχει ως συνέπεια να μην υπάρχει επαρκής προσωπικό για να μπορέσει να διασφαλίσει τον έλεγχο, παρακολούθηση των δράσεων που θα χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του ΙΠΑ. Ευχαριστώ την προσοχή σας λοιπόν στο ενδεχόμενο αυτό. Αρκούμε σε αυτά κυρία Πρόεδρε, αν έχετε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ. Η κυρία Ράουνερ της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Δάφνη, γνωρίζετε ότι είναι πολύ επιτυχημένο ε, και αγαπητό και σε αυτή την επιτροπή και στις άλλες επιτροπές ε, και χαίρομαι που θέλετε να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα, το ε, του ΣΑΕΔΑΦΝΗ γιατί πραγματικά ε, έχει περισσότερη χρησιμότητα, περισσότερη αξία για την κοινωνία, ειδικότερα τις γυναίκες καθώς υπάρχει περισσότερη προστασία, υπάρχουν περισσότερα προληπτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται μέσω αυτών των προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του Συμβουλίου, ουσιαστικά δεν υπήρξαν μεγάλε αποκλήσει από τα όσα είχε ε, προτείνει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά δηλαδή τον ετήσιο ε, σχεδιασμό, τον ετήσιο προπολογισμό. Ε, απλά υπάρχει μια πρόταση για αύξηση των ε, υποχρεώσεων κατά 350.000 ευρώ, οπότε δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή αν αξιοποιείται αναξιοποιητές επιστώσει. Δεν βλέπουμε λοιπόν προς το παρόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα του προπολογισμού σε Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μήπως η κυρία Τόμσον θα ήθελε να πει λίγα λόγια. Då är vi framme vid eh, Φαίνεται πως δεν θέλει η κυρία Τόμψο να λάβει το λόγο. Δυστυχώς έχει διακοπές το μικρόφωνο της Πρόεδρου. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διαταξή μας. Μένει να πω κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Στις 20 Εβδόμου λίγη η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Ψηφίζουμε στις 2 Σεπτεμβρίου και νομίζουμε ότι μπορούμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό ως ε, χρονοδιάγραμμα και ε, για να κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία το πρώτο αυτό εξάμεινο του έτους δουλέψατε με ενθουσιασμό και για μένα ήταν μεγάλη ικανοποίηση που μπόρεσα να συνεργαστώ με όλες και όλους εσάς. Ευχαριστώ και το προσωπικό, την Σαμπίνε, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες και συνεργάτηδες της Γραμματείας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση σήμερα. Εύχομαι σε όλες σας καλές και ξεκούραστες διακοπές. Καλό καλοκαίρι και ελπίζω όλες να μπορέσετε να αναπαυθείτε ώστε να τα ξαναπούμε τον Σεπτέμβρη όπου θα μπορέσω να σας καλωσορίσω και πάλι για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας προς επίτευξη των κοινών μας στόχων. Βέβαια, δεν μπορείτε όλες να καταλήψετε την αίθουσα τώρα. Θα παρακαλέσω να αρχίσει αμέσως η συνεδρία των συντονιστών. Που θα αρχίσει αμέσως τώρα, στις 5 η ώρα και στις 5.30.